Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψουν νέες νομοθετικές πράξεις. Σύμφωνα με την κανονική διαδικασία έχουν εγκριθεί αυτές οι νομοθετικές πράξεις.